Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Κυρίες και κύριοι, τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν καθόλου ενστάσεις. Εάν όχι, εγκρίνονται.